Mes chers collègues, un peu de silence. Λίγη ησυχία παρακαλώ. Άρχεται η συνεδρίαση. Έχετε δει την ημερήσια διάταξη. Αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις, εγκρίνεται. Οπότε, το μόνο μας θέμα είναι η τελική ψηφοφορία της έκθεσης της Επιτροπής ΤΑΞ 2. Και θα είναι η τελική μας συνεδρίαση και μετά θα έχουμε μια φιλική δεξίωση για να εορτάσουμε ε, την κατάληξη των εργασιών για το θέμα αυτό στο επίπεδό μας. Επειδή θα ψηφίσουμε, σας παρακαλώ να ελέγξετε ότι έχετε τις κάρτες σας και θα κάνουμε μια τεχνική ψηφοφορία μετά, μια δοκιμαστική ψηφοφορία για να βεβαιωθούμε ότι λειτουργούν όλες οι κάρτες και δεν υπάρχουν παραπάνω του ΕΛΚ μεταξύ των μέλων. Κύριε Πρόεδρε, υπάρχουν πάντα υπερβολικά πολλοί του ΕΛΚ, λέει ο κύριος Λαμπέρ. Ε, Ο πρόεδρος των Πρασίνων δεν έχει το λόγο. Η συνεδρίαση μας είναι δημόσια και φυσικά ε, μεταδίδεται μέσω web streaming, ως web streaming όπως οι προηγούμενες. Πρώτα απ' όλα πρέπει να εγκρίνουμε τα πρακτικά της συνεδρίας της 24 Μαΐου, αν δεν υπάρχουν παρατηρήσεις με το τέλος της συνεδρίας θεωρείται εγκρίθηκε και τα πρακτικά της δικής μας συνεδρίασης θα υποβληθούν σε διαδικασία γραπτής έγκρισης. Οπότε... Τώρα για την ψηφοφορία. Θα ελέγξουμε ότι λειτουργούν όλα σωστά. Λοιπόν, σας παρακαλώ να κάνουμε μια δοκιμαστική ψηφοφορία. Ω, Πέτερ. Πέτερ. Μήπως ένας βοηθός της ελληνικής ομάδας μπορεί να πάει να ψάξει την κάρτα σας. Α, την ξεχάσατε στην ΕΚΟΝ. Θα μπορούσε κάποιος να σας τη φέρει. Παρακαλώ. Ωραία. 39, 39, ωραία. Εκτός από τον Πέντερ, όλοι οι άλλοι, εντάξει. Πόσοι από πλευρά ΣΕΛΚ ακριβώς όσοι πρέπει, συμπεριλαμβανομένου και του εαυτού μου. Μα πρέπει να μπορέσω να ψηφίσω. Ως ΕΛΚ, όχι ως πρόεδρος. Λοιπόν, θέλω να συγχαρώ τους δύο συνεισηγητές μας, τους Κιώδης και τη Γραμματεία που έκαναν θαυμάσια δουλειά. την οποία τώρα θα υποβάλουμε στην έγκρισή μας. Τροπολογία 164 λοιπόν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 165, τις οποίες μου συντάκτη την ε, απέσυρα, για να κερδίσουμε χρόνο. 166, Dodge, υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 167, Lambert, υπέρ, κατά, αποχές, α, έλεγχος. Ελέγχουμε την 167 και θα συμμετάσχω στην ψηφοφορία. Άρχεται λοιπόν. Πέρας, πέρας. 23 υπέρ, 14 κατά, 15 κατά και δεν υπάρχουν αποχές. Εγκρίνεται. 168 Λάμπερτς υπέρ κατά αποχές δεν είναι ίδια, ο ίδιος συσχετισμός οπότε παρακαλώ να ελέγξουμε άρχεται Πέρας. 22 υπέρ, 17 κατά, μία αποχή, εγκρίνεται. 171, Λαμπέρτ, υπέρ παρακαλώ. Κατά. Και πάλι ο συσχετισμός δεν είναι ο ίδιος και πάλι ελέγχουμε, άρχεται. Είμαστε 40 πλέον. Ψηφίστε όσοι μπορείτε. Έχουμε ένα ΕΛΚ παραπάνω. Βγάζω την κάρτα μου. 39. Ψηφίσατε όλοι. Πέρας. Είκοσι υπέρ. 20 κατά. Απορρίπτεται. 170 υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα, συμβαστική 1. Υπέρ παρακαλώ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 175 Λαμπέρτς ως προσθήκη στο συμβασμό 1 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά καλά άρχεται Εγώ δεν ψηφίζω, πέρας. 21 υπέρ, 19 κατά, γκρίνεται. Οι υπόλοιπε έχουν συμπεριληφθεί και περνάμε στην 169. Ο συγητής είναι κατά υπέρ, παρακαλώ. Κατά αποχές Καλύτερα να ελέγξουμε. Εγώ δεν ψηφίζω. Άρχεται. Ψηφίστε, ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 23 υπέρ, 24 υπέρ, 17 κατά, εγκρίνεται. Συμβαστική 2 υπέρ παρακαλώ. Κατά. Α, το πρώτο τμήμα της 2 υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται επίσης. Με διαφορετικό συσχετισμό 5.44 Ρέγνερ Α, όχι, με συγχωρείτε, πίπτη. Οπότε περνάμε στη 2.51 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές Έλεγχος. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 17 υπέρ, 18, 22 κατά. Α, έχει την κάρτα τώρα. Ωραία, 17, 22 κατά, μία αποχή απορρίπτεται. Συμβαστική 3. Πρώτο τμήμα. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Το δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Επίσης εγκρίνεται. Οπότε περνάμε στην 200. Χίμπνερ. Ως προσθήκη. Υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2.15 Όχι τα σαφές. 2.15 ως προσθήκη στο συμβαστική 3 επίσης. Λοιπόν, ε, με βάση αυτά που μου λέει η γραμματεία δεν καταπίπτει το 2.15 εκτός αν ο, ο συντάκτης, ο εισηγητής θεωρεί ότι καταπίπτει. Αλλά όχι. Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. απορρίπτε νομίζω αλλά ας ελέγξουμε. Επί της 2.15. Ψηφίστε παρακαλώ. 37, 38 δεν είναι αρκετή. Α, 40. Πέρας. Ισοψηφία. 20 προς 20 απορρίπτεται. Και οι δύο του Μάρκο απορρίφθηκαν. Ε, συμβαστική 4. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 5. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Καταπίπτει 2.19. 2.16. Φίλιπ Λάμπερτσε υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Ας γίνει έλεγχος. του ψηφοφορία. παίζει η Γαλλία γιατί βλέπω ότι έχετε αρχίσει να τραγουδάτε. 20 pour. 20 υπέρ 19 κατά. Δεν, το, δεν είχα δει καλά. Δίκιο είχατε. Ζητώ συγγνώμη. 2.17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 2.18 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 2.20 ε, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται συμβαστική τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται μου λένε οι 2.34 του Λάμπερτς είναι συμβατή αντίθετα με αυτά που είχαμε πει Ω προσθήκη είναι συμβατή. Εκτό αν ε, οι συνεισηγητέ μου πούνε ότι δεν ε, το βλέπουν έτσι. Όχι, ωραία. 2.34, δεν ψηφίσουμε λοιπόν. Α, δεν ψηφίσαμε τη συμβαστική 7. Ζητώ συγγνώμη. Συμβαστική 7. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίθηκε. Τώρα η 234 είπαμε είναι συμβατή ως προσθήκη με τη συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίστε παρακαλώ. 40-41. Πολλαπλασιαζόμαστε. Φτάσουμε και τους 100. 22 προς 19. Εγκρίνεται. Συμβαστική 8 πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα είναι μια προφορική τροπολογία του ΕΛΚ. Ε, ok. partie. Τρίτο τμήμα. Wrongful or. I was wrong. Έκανα λάθος. Είπε κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τώρα η προφορική τροπολογία του ΕΛΚΠΕΡ Κατά. Έλεγχος. Μηδενίζω. 41, ωραία, πέρας. 19 προς 21 είναι η ψήφια, απορρίπτεται με μία αποχή. Η 2.37 της Ντανούτα Χιούμπνερ μπορεί να ψηφιστεί ως προσθήκη ε, για τη συμβαστική 8 που μόλις εγκρίναμε. Υπέρ. Κατά. Αποχές, έλεγχος. 39 Έχουμε επιταχύνει πάντως. Συγχαρητήρια, τα καταφέραμε. 17 προς 23, μια αποχή, ε, απορρίπτεται. Συμβαστική 9. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 2.49 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. 20 προς 19 ψήφι, δύο αποχές εγκρίνεται. 2.50 υπέρ. Κατά. Αποχές. Με τον ίδιο αριθμό ε, ψήφων εγκρίνεται. Ε, καταπίπτει 2.52, 2.53 υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Ψηφίζουμε για την 253. Ψηφίστε. 42 23 ε, ψήφι προς 16 εγκρίνεται. 2,54 είπε. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 2,55. Τη κόρα. Υπέρ. Ποιος είναι υπέρ της κόρα. Ε, κατά. Απορρίπτεται. 2.56 της Καταλήν. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Γιατί αυτή την περίπτωση πάμε στη συμβαστική 10. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται επίση με λίγο διαφορετικό αριθμό ψήφων. 2,88 καταπίπτει. 2,74 του Γκούναρ Χέκμαρ υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 11. Συμβαστική 11 δηλαδή. Πρώτο τμήμα. Κατά. Η είναι κατά. Το χέρι της υπερβόνωση ε, λέει όχι, αλλά το στόμα της ναι. Θεωρήσουμε ότι είναι κατάφαση η απάντηση. Λοιπόν, ε, δεύτερο τμήμα τώρα, υπέρ, κατά, αποχές, γιατί άλλαξε ο τρόπος που ψηφίσατε, οπότε νομίζω ότι εγκρίνεται. Έλα, μην, τα, μην, εγκατα, εγκαταλείπετε. 41-42. 25 προς 16. Μία αποχή εγκρίνεται. Ε, τρίτο του. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τμήμα 4, όχι 2, ξαναλέει 2. Τμήμα 4, λοιπόν, πάλι το wrongful. Ποιο είναι υπέρ του wrongful, κατά. Αποχές, κανείς δεν σηκώνει πλέον τα χέρια του. ψηφιστε 40-41-42 πέρας, 27 προς 14, μία αποχή εγκρίθηκε. Ε, άρα, μόλις εγκρίναμε συμβαστική 11, ε, ήδη προσθήκης 2.84. Ε, Ποιος είναι υπέρ της 2.84, κατά. Ε, δεν υπάρχει μεγάλη διαφορά, οπότε χρειάζεται να κάνουμε έλεγχο. Ψηφίστε παρακαλώ. Α, ισοψηφία 21 προς 21. Η ψήφη απορρίπτεται, Ντανούτα. 2,79. Άλλη προσθήκη από τον Φίλιπ Λάμπερτ. Αυτή τη φορά υπέρ. Κατά. Απόχες. Νομίζω ότι απορρίπτεται. Θα ελέγξουμε. Για λόγους πολιτικής συμμετρίας και ισορροπίας ψηφίστε 41-42 πέρας. 20 προς 21. Μία αποχή απορρίπτεται. Έτσι, Φτάσαμε στη 287 Τον ε, Φερνάντες και Χάουρεγγια Τόντο. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική 12. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται επίσης αυτό μας επιτρέπει να ψηφίσουμε τώρα συμβαστική 13 ομού. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίθηκε. Στην 309 φτάνουμε τώρα, Φίλιπ Λάμπερτς. Υπέρ, κατά. Απόχες. Έλεγχος, παρακαλώ ψηφίστε. 41 ψήφισαν, 21 ψήφοι υπέρ, 20 κατά, εγκρίθηκε με διαφορά μιας ψήφου. 3-10, Πολ Τάγκ, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβαστική 14, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, είναι προσθήκης και πάλι. Φίλιπ Λάμπερτ, 3-15, υπέρ κατά και πάλι μικρή είναι η διαφορά. Νομίζω ότι μάλλον απορρίπτεται. Θα το εξακριβώσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Γρήγορα παρακαλώ. Προχωρούμε πολύ γρήγορα. 21 ε, ψήφοι προς 21 αποχή εγκρίνεται. Σύμβαστηκε 15. Σε τρία τμήματα λέει ο πρόεδρος. Όχι, όχι, αυτά είναι στη, για τη 16. Δεν βλέπω καλά σήμερα. Συμβαστική 15 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ε, η συμβαστική 16 είναι που είναι χωρισμένη σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, binding union υπέρ, κατά. CR, έτσι, εποχέ εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, Εξακριβώ. Ψηφίστε για το τρίτο τμήμα της συμβαστικής 16. Ένας ε, από τους πρασίνους. Ε, απίστευτο μου φαίνεται. Πού είναι η πράσινη. Ποιος είναι. Εκτό και αν ήρθε κάποιο καινούριο στην ομάδα, εγώ πάντω δεν το ξέρω. πώ είναι η τεχνητή νοημοσύνη, ένα υπολογιστή. Όχι, γιατί η δική μα δεν είναι τεχνητή ευθεία, είναι πραγματική, απαντάει ο κ. Λάμπερτ. Υπάρχει μια πράσινη κάρτα ψηφοφορία ε, ή κα, κάποιος έχει ε, διχασμένη προσωπικότητα, δεν ξέρω, σε εμά δεν νομίζω, υπερβάζουμε, γιατί μας λέγατε πριν ότι άλλα λέει το χέρι της, άλλα λέει το στόμα της για αυτή τη διγλωσία και είπαμε πως έχει διχαστεί. Σταματάμε την, ε, διακόπτουμε την ψηφοφορία. Την ακυρώνουμε και την επαναλαμβάνουμε. Ψηφίζουμε και πάλι. μαγεία. Είναι η 43η ψήφος. Είναι ε, μία παραπάνω από ό,τι πρέπει. Δεν γίνεται αυτό. Είναι... Α, α 42 ψήφισαν. 43 είναι αλλά 42 ψήφισαν. Να την ναι. Του Φερνάντε τι θέση ήταν. Λοιπόν, καλά. 42 ε, ε, οι ψηφίσαντε, 42 οι κάρτε. Ε, κανένα πρόβλημα. Μα ε, το μηχάνημα λέει ότι έχουμε ένα πράσινο παραπάνω, όχι σοσιαλιστή. Τέλο, πάντων, τι λέει το, το αποτέλεσμα. 25 ψήφοι προς 17 εγκρίνεται. Αυτό ήταν το τρίτο τμήμα. Περνούμε στην 326, πάλι ε, είναι προσθήκη για τη συμβαστική 16, ε, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτω. Μην ε, ξαναπολαπλασιαστούν τώρα οι πράσινοι ξαφνικά. Είναι ένας πράσινος παραπάνω. Δεν καταλαβαίνω. 21 ψήφους 19, δύο αποχές. C'est quand même un mystère. Comment Τι να κάνουμε τώρα, δεν αλλάζει τίποτα σε αυτή την ψηφοφορία. Non, ça change pas ce vote, même si on enlève 21 moins 1. 21 ψήφοι, μείον αυτή την ψήφο, 20. Πάλι δεν αλλάζει η έκβαση ψηφοφορίας. Συγγνώμη, 21, ε, ε, ε, όλα δεν, δεν δεν ε, ε, σας δίνω το λόγο γιατί μόνο τα μέλη της Επιτροπής όταν τους δώσει ο πρόεδρος το λόγο τότε μπορούν να μιλήσουν. Πρέπει να το λύσουμε αυτό το πρόβλημα οριστικά. Τι είναι αυτή η κάρτα εκεί πέρα μόνη της. Πιανού κάρτα είναι αυτή. Είναι δική μου η κάρτα. Εσείς δεν είστε πράσινοι. Η FTD είμαι. Το Μάρκο Βάντι καθιστώ. Μπορείς να αλλάξετε να καθίσετε δίπλα. Συγγνώμη, Πρόεδρε, το να αλλάξει κάθισμα δεν σημαίνει ότι αλλάζει κάτι στο μηχάνημα τη ψηφοφορία. Α δούμε παρόλα αυτά, λέω. 17, υπέρ. Κατά. Απόχες. Εγκρίνεται. 3.36. Υπέρ. Κατά. Απόχες. Απορρίπτεται. Συμβαστική η 18 υπέρ, σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά. Απόχες. εγκρίνονται Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα ελέγξουμε. Θα δούμε αν ε, η αλλαγή καθίσματος αλλάζει κάτι στη, στο αποτέλεσμα. Oui, c'est la magie 37 ça va, 38 ça va, ça y est. Au 39, bon. 39 ψήφισαν. Για να είστε παρακαλώ, για να εξακριβώσουμε τι έχει συμβαίνει. Έχουμε 25 εδώ υπέρ, 16 ε, κατά και καμία αποχή, έτσι. Θα κάνουμε μία έξα ακριβώς, σήκω στα χέρια. Υπέρ. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, δεν 25.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 Είναι αρκετά διασκεδαστική η κατάσταση. Διανάταση χειρός εξακριβώνουμε αν έχει κάνει λάθος ή όχι το μηχάνημα. Είναι δημιουργικός τρόπος στην ψηφιακή εποχή. Αυτό ήταν το πρώτο τμήμα. Ε. το δεύτερο. Τρίτο τμήμα ε, της συμβαστικής 18. Υπέρ. Κατά. Έλεγχος. Φιλίπ, είστε υπέρ ή κατά. Αφού λειτουργεί καλά το μηχάνημα, όπως μόλις διαπιστώσαμε, ψηφίζουμε ηλεκτρονικά για το τρίτο τμήμα της συμβαστικής 18. Συγκλονίζεται και πάλι το μηχάνημα. 25 προς 17. Εγκρίνεται. 3.48. Μπεντ Λούκε δυστυχώ δεν μπορείς να έρθει. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η συμβαστική 19. Μπλοκ. Ε, υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 3.48 του Λούκε. Υπέρ κατά δύο φορέ σήκω στο χέρι του Φίλιπ Λάμπερτ. έλεγχο. 3.48 του Μπεν Λούκε Ξακολουθεί να κάνει τρελά το μηχάνημα 42 Ωραία 26 προς 16 αποχές εγκρίνεται. Ε, συμβαστική 21ο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά αποχές ελέγχος. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας 23 προς 17, δύο αποχές εγκρίνεται και καταπίπτει 3.55 συμβαστική 21 σε τρία τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ. Κατά. Αποχές. Ελεγχός. Ψηφίστε για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής τροπολογίας 21. Le vote est clos. 25 pour 17. 25 υπέρ 17 κατά η ίδια πλειοψηφία εγκρίνεται. Τρίτο τμήμα της, ε, της ε, πρότασης αυτής υπέρ κατά εγκρίνεται ολόκληρη η σημαστική εγκρίνεται πράγμα που σημαίνει ότι πάμε στην 364 πολτάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. αν δεχτούμε ότι ο Φίλιπ Λαμπέρτ ψήφισε υπέρ. Συμβαστική 22 σε δύο τμήματα. Πρώτο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η 371 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 372 Απορρίπτεται η 371. 372 της κόρα. Υπέρ. Κόρα. <laughs> Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Μεγάλη, απόλυτη μοναξιά της κόρα. Δεύτερη ευκαιρία. 374. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Όχι. Πάλι όχι. Δεν είναι η βραδιά σας απόψε κόρα. 373. Φιλίπ Λαμπέρτς. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 375. Τόμ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Η 376. Φιλίπ Λαμπέρτς. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία για την 376. Ψηφίστε παρακαλώ. 42, 40 ψήφισαν. Πέρας, 22 υπέρ 18 κατά, δεν υπάρχουν αποχές, εγκρίνεται. 377 του ιδίου. Υπέρ, κατά, αποχές, η ίδια πλειοψηφία, εγκρίνεται. 378 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 379 του ιδίου υπέρ κατά αποχές με την ίδια πλειοψηφία. Εγκρίνεται. Συμβαστική 23, πρώτο τμήμα, υπέρ. Κατά. Ένας από τους συνεισηγητές είναι κατά. Α, ήταν λάθος, μάλιστα σε, κόλλησα στην ασθένεια του Φιλίπ Λαμπέρτς. Κι εγώ εξάλλου. Κύριε Πρόεδρε, δεν είμαι <laughs> άρρωστος. Έχω πιει, λέει ο κύριος Λαμπέρτς. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Πάμε στην συμβαστική 24 και πάλι σε δύο τμήματα. Ε, πρώτο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία υπέρ, αλλά στο ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίζουν όλοι. Είμαστε 41 μόνο τώρα. 25, 16. Δεν υπάρχουν αποχές. Εγκρίνεται. Περνάμε την 547 ως προσθήκη στην 24. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται με την ίδια πλειοψηφία. Συμβαστική 25. Υπέρ, α, συγγνώμη, πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, αποχές, Νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία, αλλά ας το ελέγξουμε. Ας το επαληθεύσουμε. Ψηφίστε όμως, ε, γιατί κάποιοι αποκοιμήθηκαν. 38 δεν είναι ικανοποιητικό. 41. 26 υπέρ, 15 κατά. Δεν υπάρχουν αποχές, εγκρίνεται. Οι 394 λοιπόν καταπίπτει. Συμβαστική 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Στην 397, 398 ε, με συγχωρείτε Δανούτα, υπέρ. Η Δανούτα είναι υπέρ, αλλά είναι η μόνη. Κατά. Όσοι δεν είναι ΕΛΚ είναι κατά. Αποχές. Έχει απομονωθεί το ΕΛΚ. Είπατε ότι όσοι δεν είναι έλικα, αλλά όσοι είναι. Αυτή, αυτή η παρατήρηση είναι απαράδεκτη, ακόμα και ως χιουμοριστική. Η Ντανούτα λοιπόν έχει στεναρή υποστήριξη της ομάδας της, αλλά είναι απομονωμένη στην Επιτροπή μας. 399. Άννα Γκόμες, υπέρ, κατά. Αποχές. Θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Λείπουν ακόμα μερικοί. Πέρας. 20 υπέρ, 19 κατά μία αποχή. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική τροπολογία 27. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Ερχόμαστε έτσι στην 408 τον 2 Μάρκο. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 409. Φίλιπ Λεμπέρτς, Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 411. Αλέλα Μασούρ. Υπέρ. Ποιος τολμάει να είναι κατά. Αποχές. Η πιο σημαντική ψηφοφορία της βραδιάς. Εγκρίνεται. 419 του Φάμπιο. Υπέρ, κατά, αποχές. Νομίζω ότι υπάρχει πλειοψηφία υπέρ, αλλά στο ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας. 21-19 μία αποχή εγκρίνεται. Συμβιβαστική 28. Πρώτο τμήμα. Ψήφι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές το ΕΛΚ λοιπόν εδώ εγκρίνεται. Κάποιος ζητάει έλεγχο ηλεκτρονικό για το δεύτερο τμήμα της συμβαστικής 28. Ψηφίζουμε για το παράρτημα. Φορά το παράρτημα. Πέρα τη ψηφοφορίας. 24 υπέρ, 2 κατά 15 εποχές. Εντάξει. Λοιπόν, αποφασίζουμε να βάλουμε στο παράρτημα το κείμενο των φίλων μας πρασίνων. Και θα δημοσιευθεί αφού ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία. Ε, 419. Φάμπιο και Σβέν. Ως προσθήκη στην 28. Υπέρ, κατά, αποχές, θα το ελέγξουμε ευθύ αμέσω. Για την 419. Ψηφίζουμε. Πέρας. 21, 19, μία αποχή. Εγκρίνεται. 443 των ιδίων και πάλι ως προσθήκη υπέρ, κατά, αποχές, υπάρχει η ίδια πλειοψηφία. Καταπίπτει 444, 410 επίσης. Ψηφίζουμε την 425 των πρασίνων. Υπέρ, κατά, αποχές, πρέπει να το ελέγξουμε. Είναι πολύ κοντά το αποτέλεσμα. Ας ψηφίσουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Λείπει μία ψήφος. Πέρα της ψηφοφορίας. 22 υπέρ 19 κατά. Εγκρίνεται. 426 υπέρ. Κατά αποχές θα το ελέγξουμε και αυτό το αποτέλεσμα. Είναι δύσκολο γιατί δεν σηκώνετε όλοι τα χέρια σας. Για την 426 λοιπόν. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 22 υπέρ, 19 κατά. Η ίδια βιβλιοψηφία 427. Εδώ θα είναι διαφορετική η πλειοψηφία. Υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται. Συμβιβαστική 29. Ψήφι υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 436 Φάμπιο και Σβέν υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε. Νομίζω ότι υπάρχει μια μικρή πλειοψηφία. Άρχεται η ψηφοφορία, Υπέ... Ε, ψηφίσατε όλοι, πέρας. Α, όχι, κάτι έγινε εδώ, δεν μπορεί. 34 υπέρ και 7 κατά. Η όρασή μου κάτι έχει σίγουρα. Αυτή ήταν η 436, 437 υπέρ. Κατά, αποχές, εδώ αξίζει να το επαληθεύσουμε για την 437. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 22 υπέρ, 19 κατά. 0 αποχή. Αποχές. Η άλλη καταπίπτει. Πάμε στην 446. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 447. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 448 θα πρέπει να τεθεί σε ψηφοφορία. Λοιπόν, υπέρ κατά αποχές θα το ελέγξουμε για την 448 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 17 υπέρ 20 κατά 4 εποχές απορρίπτεται 449 της Καταλήν υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται θα το ελέγξουμε. Νομίζω ότι υπάρχει ο ίδιος σχετισμός, αλλά θα το ελέγξουμε αφού θέλετε. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 17 υπέρ 19 κατά 4 εποχές όντως απορρίπτεται. 450. Πρέπει να ψηφίσω, λέει ο πρόεδρος. θα, αλλάξουν τα πάντα. 450 του Μπράιαν. Υπέρ. Κατά. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική 30. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα το ελέγξουμε. Και έτσι ψηφίζω και εγώ. Για το δεύτερο τμήμα είναι οι οδηγίε του ΕΛΚ. Άρχεται η ψηφοφορία. 24 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Πράγμα το οποίο μας φέρνει στην συμβαστική τροπολογία 31. Τμήμα 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα υπέρ κατά, αποχές, θα το ελέγξουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. Το έλκα από ό,τι καταλαβαίνω ψηφίζει κατά. 20 υπέρ, 19 κατά, 3 αποχές, εγκρίνεται και το δεύτερο τμήμα. Έτσι ερχόμαστε στην ε, τροπολογία 463 της Σιλβί Γκουλάρ και Νίλς Τόρβαλτς. Υπέρ. Κατά. Αποχές θα το ελέγξουμε. Για την 463. Σιλβί Γκουλάρ, Νίλς Τόρβαλτς. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 19 υπέρ, 20 κατά, 3 αποχές. Απορρίπτεται άρα. 464 αναγόμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 465 ντανούτα που είναι συμβατή υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβιβαστική 32 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές και αυτό εγκρίνεται. Με μικρότερη πλειοψηφία, αλλά εγκρίνεται. Έτσι ερχόμαστε στην τροπολογία 477 των συνεισηγητών, που δεν είναι όμως συμβαστική. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 474, υπέρ, κατά, αποχές, Εγκρίνεται. Νομίζω, καταλαβαίνω ότι το ΕΛΚ είναι κατά. 475 υπέρ, κατά, αποχές. Ας γίνει έλεγχος. Προσπαθείτε να σηκώνετε το χέρι σας. Για την 475 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Κάποιο δεν έχει ψηφίσει ακόμα. Εντάξει. 21 υπέρ 19 κατά δύο αποχέ, Εγκρίνεται. Συμβιβαστική 33. Πρώτο τμήμα. Υπέρ. Κατά. αποχέ, Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Από έχουν οι πράσινοι. Άρα θα πρέπει να το επαληθεύσουμε το αποτέλεσμα για το δεύτερο τμήμα της 33. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πρέπει να ψηφίσω κι εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Ψηφίστε παρακαλώ. 23 ψηφίοι υπέρ, 16 κατά, 3 αποχές εγκρίνεται. 480 ως προσθήκη στην 33 το Φίλιπ Λαμπέζ. Υπέρ, κατά, αποχές το ελέγξουμε. θα το ελέγξουμε. Η 480 τροπολογία ψηφίζουμε 41, λείπει ο 42 22 υπέρ, 18 κατά, 2 αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 34. Πρώτο τμήμα, ψήφι υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Έρχομαστε έτσι στην 488 που ζητάει διαγραφή. Υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 489 των εισηγητών. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. <laughs> Δυστυχώ, η 466 καταπίπτει. Κατά τον τρόπο αυτό, ομόφωνα εκφράζουμε τη λύπη μας. Πάμε στην 490. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβαστική 35. Πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχέ, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Για απελυφή τη λέξη public. public. Υπέρ, κατά, αποχές, θα το ελέγξουμε, πιστεύω ότι υπάρχει πλειοψηφία. Αλλά επειδή είναι τόσο σημαντική αυτή η λέξη, ψηφίζουμε πέρα της ψηφοφορίας, 24 υπέρ 17 κατά μία αποχή, το public εγκρίνεται. Αυτό μας φέρνει στην τροπολογία 36, τη συμβιβαστική. Ε, υπέρ κατά, το ΕΛΚ είναι κατά. Θα ελέγξουμε λοιπόν το αποτέλεσμα για την Συμβαστική 36, έτσι δεν είναι. Η 36. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 21 υπέρ, 17 κατά, 4 εποχές, η 36 εγκρίνεται. Η 37. Πρώτο τμήμα. Η 280 δεν εγκρίθηκε, έτσι δεν είναι. Άρα ψηφίζουμε για την 37, το πρώτο τμήμα. Υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα, υπέρ, κατά, ε, έλεγχο ηλεκτρονικό, το δεύτερο τμήμα νομίζω ότι εγκρίθηκε, αλλά προτιμώ προτιμώ να το ελέγξουμε. 42 ε, ψήφισαν, 20 προς 19, τρεις αποχές, εγκρίνεται. Justesse. Et... Ε, Οπότε, να δούμε τώρα το τρίτο τμήμα για το TTIP υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. Οπότε, μα οι δύο μεγάλες ομάδες καταψήφισαν. Α, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις. Δεν ξέρω αν και εγώ έχω διαφορετικές απόψεις για το θέμα αυτό. Το ΕΛΚ, ε, στο ΕΛΚ υπάρχουν ε, διχογνωμίες επ' αυτού. Εν να ελέγξουμε το τρίτο τμήμα της συμβαστικής 37. Ψηφίστε παρακαλώ, ψηφίστε. Ψηφίστε είτε έτσι είτε αλλιώς, αλλά ψηφίστε. Πέρας. 15 υπέρ, 26 κατά μία αποχή. Απορρίπτεται. Το τρίτο τμήμα. Οπότε είμαστε στην 514 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 515 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 5.16 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Βλέπω ότι ο συντάκτης δεν ψήφισε. 5.17 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 5.18 καταλήν υπέρ κατά αποχές έλεγχος της 5.17 άρχεται. Ψηφίστε παρακαλώ, ψηφίστε. Πέρας. 21 ψήφι, ισοψηφία, υπέρ και κατά, απορρίπτεται. 5-19 υπέρ. Κατά. Αποχές. Καλύτερα να ελέγξουμε. Γιατί δεν βλέπω να σηκώνετε τα χέρια σας. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε πέρας. 22 υπέρ 20 κατά. Εγκρίνεται. 5.20 υπέρ κατά αποχές ίδιος συσχετισμός εγκρίνεται 5.21 Χακμαρχ υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι απορρίπτεται αλλά ελέγχουμε την 5-21. γιατί είναι πολύ ε, αμφίροπα αυτά τα αποτελέσματα. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 19 υπέρ, 22 κατά, μία αποχή, απορρίπτεται. 5-22 του ιδίου υπέρ. Κατά. Με ευρία πλειοψηφία απορρίπτεται. Συμβαστική 38 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 5-23 ως προσθήκη στην 38. Μαρκοτζάνη Μαρκοβάλι, Υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Περνάμε τώρα στην 5.33. Λαμπέρτς υπέρ. Κατά αποχές. Το έλκτη δεν καταλαβαίνω. Το ΕΛΚ δεν καταλαβαίνω τι ψηφίζει. Εν πάση περιπτώσει, ας ελέγξουμε. 5.33. Και στο το ΕΛΚ συμφωνεί υπάρχουν οικονομίες. Για να ξέρω τι θα κάνω κι εγώ. Θα χωριστώ στα δύο. 22 υπέρ 20 κατά. Εγκρίνεται. 5.34 υπέρ. Οι σοσιαλιστές, οι δεν είναι υπέρ. Κατά παρακαλώ ποιοι είναι. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Γιατί βλέπω ότι κάποιες μεγάλες ομάδες ε, ψηφίζουν προς δύο διαφορετικές κατευθύνσεις. Ψηφίστε παρακαλώ, ψηφίστε. Ψηφίστε παρακαλώ προς τη μία ή την άλλη κατεύθυνση. Πέρας. 23 υπέρ 18 κατά εγκρίνεται. Χάρη στο ΕΒΚΙ 535 υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε και πάλι. Γιατί βλέπω ότι οι ορισμένε ομάδες ψηφίζουν διαφορετικά από την προηγούμενη φορά. Ψηφίστε πέρας. πέρα. Λοιπόν, τώρα απορρίπτεται. 17-24 μία αποχή απορρίπτεται 5.35 περνάμε στην 5.36 υπέρ κατά να την ελέγξουμε και αυτήν 5.36 έχουμε τέσσερις τροπολογίες των ιδίων 5.36 ψηφίσατε όλοι πέρας 17 υπέρ 24 κατά μία αποχή απορρίπτεται και τέλος η 5.37 υπέρ κατά αποχές να ελέγξουμε και αυτήν νομίζω ότι είναι ίδιος ο συσχετισμός αλλά επειδή είναι αμφίροπα τα αποτελέσματα ας ελέγξουμε 16 υπέρ 25 κατά μία αποχή απορρίπτεται 5.38 Ντανούτα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η 539 δυστυχώς έχει αποσυρθεί από τον συντάκτη της. Ε, παραρτήματα. Παράρτημα 1. Μια τεχνική τροπολογία. Συμφωνούμε όλοι, εντάξει. Ωραία. Για το δεύτερο παράρτημα. Το λάβουμε υπόψη στη συμβαστική 28. Παραρτήματα 3α έως 3b4 έχουμε την τροπολογία 540 Το πρασίνο, Ποιοι είναι υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές εγκρίνονται. 541 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Περνάμε στις ιδεολογικές σκέψεις. Τροπολογία 11 των πρασίνων υπέρ παρακαλώ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Την 11 άρχεται. Ψηφίστε, ψηφίστε. Ψηφίστε. Πέρας. Με 21 ψήφους υπέρ και 20 κατά και μία αποχή εγκρίνεται. 12 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 13 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 14 των ιδίων υπέρ. Κατά. Αποχές το, αυτό αποτέλεσμα. Συμβαστική 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ. Κατά. Αποχές έλεγχος. Της 21. Άρχεται. Πέρας. 20 υπέρ, 22 κατά, μηδεν αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 22 υπέρ κατά αποχές ορισμένοι ήταν διστακτικοί οπότε ας ελέγξουμε την τροπολογία 22 της Ντανούτα. Ψηφίστε, ψηφίστε. Πέρας. 18 υπέρ 24 κατά απορρίπτεται. Συμβαστική 40. Συνολικά υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 30. Γκουλάρ Τόρβαλτ υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 31. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε την 31. Άρχεται πέρα Με 21 ψήφους υπέρ και 20 κατά και μία αποχή εγκρίνεται. 32 των πρασίνων υπέρ. Κατά αποχές να ελέγξουμε. Την 32 άρχεται. Συνεχίζεται, συνεχίζεται, αλλά κλείνει. 21 υπέρ, 20 κατά μία αποχή θα έπρεπε να καταψηφίσει αυτός που απέχει. Θα είχε πιο πλάκα. Εγκρίνεται. 33. Χοκμαρκ. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Την 33. Να ελέγξουμε την 33. Ποιος θέλει 33. Υπέρας. 17 υπέρ 24 κατά. Μία αποχή. Ο Γκουνάρ δεν αγοράζεται. 34 των πρασίνων. Υπέρ κατά. Οι σοσιαλιστές τι κάνουν. Είναι υπέρ. Α, κατά. Καλά κοιτάξτε θα ελέγξουμε. Γιατί δεν είναι σαφές. Ελέγχουμε την 34. Την 34. Πέρασε. 21 υπέρ 20 κατά μία αποχή. 35 υπέρ κατά καλά να ελέγξουμε γιατί γιατί και εδώ θα είναι παρόμοιο το αποτέλεσμα αλλά ένας να ψηφίσει διαφορετικά αλλάζει το αποτέλεσμα ψηφίστε παρακαλώ ψηφίστε ε, ευχαριστώ 21 πέρα 20 κατά και η μία αποχή θαυμάσια συνέπεια σε αυτές τις ε, τόσο αμφίρωπες ψήφους 36 των ιδίων. Η ίδια πλειοψηφία. Λοιπόν, να ελέγξουμε απευθεία. Θα μπορούσαμε να σας κάνουμε μία τιμή χονδρικής, λέει ο κ. Λάμπερτ. Ναι, αλλά ορισμένοι δεν ψηφίζουν ε, ακριβώς με τον ίδιο τρόπο. Δεν ψηφίζουν με βάση το συντάκτη, αλλά με βάση το περιεχόμενο. Ψηφίστε παρακαλώ. 42. πέρα. 22 υπέρ. 20 κατά. Αυτός που απήχε τελικά πέρασε με το Φιλίπ. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται με ευρία πλειοψηφία. Συμβαστική 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 των πρασίνων. Υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 43 Λούκε υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 44 Χόκμαρκ υπέρ κατά αποχές ας την ελέγξουμε αλλά νομίζω ότι έχει απορριφθεί αλλά από σεβασμό προς τον Χόκμαρκ ας ελέγξουμε αλλά παρακαλώ ψηφίστε όλοι ψηφίστε ψηφίστε ψηφίστε Πέρασε. 17 περί 24 κατά, όντως απορρίπτεται. 45, Λαμπέρτ, υπέρ. Κατά. Mm. Εδώ βλέπω ότι γίνεται άλλου τύπου παιχνίδι. Οι πράσινα υποστηρίζονται από το ΕΛΚΑ περίεργο. Ας ελέγξουμε. Ψηφίστε παρακαλώ. Ψηφίστε. Πέρας. 23 υπέρ 18 κατά μία αποχή εγκρίνεται η τροπολογία 45 καταπίπτει λοιπόν 46 47 υπέρ παρακαλώ κατά αποχές βλέπουμε αυτήν την διαφορά απόψεων αλλά πρέπει να τη μετρήσουμε ψηφίστε παρακαλώ ψηφίστε ένας ε, κουράστηκε δεν ψηφίζει πια. Πέρας. 22 υπέρ 18 κατά μία απόχη εγκρίνεται. 48 Dodge. Η νέα μητέρα. Ποιοι είναι υπέρ της νέας μητέρας. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 49 των πρασίνων. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Να ελέγξουμε. Την 49. Ελέγχουμε ναι, 49. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας. 21 μία ψήφι υπέρ, 20 κατά, μία αποχή. Είναι δύσκολα. Συμβαστική 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 53 ως προστίκη στη συμβαστική 42. Υπέρ. Κατά. Αποχές για να ελέγξουμε την, 40, την 53 τροπολογία. Σλάιν Μακάβαν. Ψηφίστε παρακαλώ. Ωραία. Πέρασε. 23 υπέρ 18 κατά μία αποχή. Εγκρίνεται. 56. Τη Σάλντε υπέρ παρακαλώ. Κατά. Αποχές. Ας ελέγξουμε. Γιατί ένα τμήμα των αριστερών δεν είναι υπέρ. Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρασε. Ναι, πρέπει να ελέγξουμε. 20, κατά, 20 πέρα, 21 κατά και μία αποχή απορρίπτεται. 57 το υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 58 μορέλ υπέρ. Κατά. Αποχές ε, νομίζω ε, θα εγκριθεί αλλά εξακρίβωση. 58. Μορέλ. Ψηφίστε παρακαλώ 22 προς 20. Εγκρίνεται. 59. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Για την 59 α, αποκλείεται να προφέρω ε, το όνομα του συντάκτη γιατί δεν θέλω να το παραθύρω. Από σεβασμό δηλαδή για τη γλώσσα του 19 προς 23 απορρίπτεται. Η 60 το υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. 61 υπέρ. Κατά. Αποχές ε, απορρίπτεται. 62 τανούτα υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται 63 της Ντανούτα υπέρ. Κατά. Αποχές ε, έλεγχος για την 63. Έλεγχος για την 63. Ψηφίστε, ψηφίστε. Πέρασε 17 προς 24, μία αποχή απορρίπτεται. 64 των πράσινων υπέρ. Κατά Αποχές απορρίπτεται. 65 το των είναι υπέρ. Κατά. Πάλι ε, συμμαχία κατά φύση. Εξακρίβως για την 65. Παραφύση, συγγνώμη, για την 65. Ψηφίστε, ψηφίστε, ψηφίστε. Πέρας. 21 ψήφοι προς 20 και εγκρίθηκε. 66 έχει αποσυρθεί. 67 των πρασινών υπέρ. Κατά. Αποχές είναι πιο φυσιολογική αυτή η συμμαχία, αλλά θέλω παρόλα αυτά να εξακριβώσω αν ισχύει. Την 67 παρακαλώ ψηφίζουμε ηλεκτρονικά. Πέρας. 23 προς 18 μια εποχή 73 70-30 νότα υπέρ... Α, καταπίπτει. Συγγνώμη, ολόκληρη σειρά των τροπολογιών μέχρι την 74. Ψηφίζουμε για την 74 πράσινη υπέρ... Κατά... Αποχές... Παρά το διχασμό του ΕΛΚ εγκρίθηκε η τροπολογία. Συμβαστική 43 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. Μπούρκαρτ Μπάλτς 77 σε, για, ως προσθήκη υπέρ. Κατά. Αποχές εξακρίβωση ευθύ αμέσω για την 77. Ψήφιστε, ψηφίστε, ψηφίστε. 23 προς 17, δύο εποχές. Εγκρίθηκε ως προσθήκη. Και έτσι πάμε στην 83. Σωστά, ναι, 83, πράσινη, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 543, υπέρ, κατά, αποχές εξακρίβωση η γνωστή διαφορά ανάμεσα στην δεξιά και την αριστερά όμως πρέπει να είμαστε πιο συγκεκριμένοι Αχα, 21 προς 20 μια αποχή ενδιαφέρον θα ήταν να δούμε ποιος ε, απέχει 84 Μορέλ υπέρ Α, όχι, καταπίπτει. Καταπίπτουν οι δύο επόμενες. Άρα περνάμε στην 87. 87 πράσινη πάλι υπέρ. Κατά. Ναι, αλλά είπαμε ότι αν εγκρίνει η 83 καταπίπτει, έτσι δεν είναι. Όχι, ζητώ συγγνώμη, μπράβο. Σωστή παρατήρηση. Την 85 αλλά και την 84 Εγκρίθηκε η 543, άρα η 84 κατέπεσε. Αντίθετα η 85 που είναι συμβατή με την 543. Πρέπει να ψηφιστεί γιατί απορρίφθη η 83. 85 λοιπόν, υπέρ. Κατά. αποχές απορρίπτεται όχι τα να είναι μού την ψηφοφορία και υπό το φοροτιμής στο συντάκτη ε, 87 ε, πράσινη υπέρ κατά αποχές Άντε πάλι διασταυρούμενες συμμαχίες, ε, πρέπει να το επαληθεύσουμε. 87 ψηφίστε, ψηφίστε. 23 προς 18, μία αποχή εγκρίθηκε. Άρα κατά καταπίπτει 86, συμβαστική 44. Τώρα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 πράσινη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται η συμβαστική 45 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται 98 του κυρίου Μονό υπέρ. Ο κ. Μονό είναι υπέρ. Είναι και κάποιο άλλο υπέρ από Έδωσε, όχι απερίφθη. 46, συγγνώμη, υπέρ κατά αποχέ. Εγκρίνεται η 104 των πράσινων υπέρ. Κατά αποχές επαλήθευση για την 104 πέρας 20 μία προς 20 μία αποχή η 105 λοιπόν θα είναι η ίδια πλειοψηφία υπέρ κατά αποχές ψηφίσατε όλοι το ίδιο όχι άρα το ίδιο αποτέλεσμα ε, συμ... Εγκρίνεται δηλαδή. Συμβαστική 47. Υπέρ. Κάτα. Αποχές ε, εγκρίνεται. 8 των πρασίνων υπέρ. Κατά. Αποχές. Επαλήθευση. Αν ενδεχομένω ε, σημειώνονται διαφορετικά αποτελέσματα ε, κάποιες φορές 23 προς 19, ε, ναι, είναι ελαφρώς διαφορετική πλειοψήφια. Λοιπόν, 109, Πολτάν. υπερκάτα απόχες, επαλήθευση για την 109. Ψηφίστε παρακαλώ για την 109. 109. Ψηφίστε, ψηφίστε, ψηφίστε. Πέρας. 22 προς 20 εγκρίνεται. Συμβαίνει 110 των πρασίνων υπέρ. Πολύ. Λαός. Κατά. Λιγότεροι. Εποχές. Εγκρίνεται. Συμβαστική 48. Μία τροπολογία έχει συμπεριλαμβάνει. Α, όχι, όχι, όχι. Πολλές. Συμβαστική 48. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίθηκε. Και στην 115 προσθέτουμε ε, σε σχέση με τη συμβαστική 48 υπέρ, κατά. υπάρχουν και ενστάσεις. Επαλήθευση, η 115 είναι προσθήκη στην συμβαστική 48. Ψηφίστε, ψηφίστε, ψηφίστε. Διατηρούμε το ρυθμό μας, ε, ορίστε 19 προς 22, μία αποχή, απορρίπτεται, δεν προστίθεται τίποτα 48, 116 νούτα, υπέρ. Απολογία 116 υπέρ, κατά. Επαλήθευση, νούτα. Πέρας. 17 μόνο προς 24 ιτήθηκε η Ντανούτα. 117 Μάρκο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Μ, το επαληθεύσουμε για το L και υποστηρίζει το EFTD. Δεν καταλαβαίνω εγώ τέτοιες λεπτές χρειές. Επαλήθευση. 117. 19 προς 22 αποχή παρά τις προσπάθειες που κάναμε αγαπητέ Μάρκο ιτήθηκες 118 της Έστερ ποιος είναι υπέρ της Έστερ α συγγνώμη πρώτα την 119 των πράσινων 119 υπέρ κατά αποχές ε, απορρίπτεται 118 της Έστερ υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 120 πράσινο πάλι υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 49 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 127 των πρασινών υπέρ κατά αποχές επαλήθευση για την 127 Ψηφίστε παρακαλώ. Πέρας 20 προς 21. Ε, Απορρίπτεται. 128 της ΓΚΟΕ Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 131 ε, ε, η ΓΚΟΕ υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 132 πράσινη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 50 ομού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 139 υπέ, επράσινη υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 138 πολτάν υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 140 πράσινη υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβαστική 51 υπέρ κατά ΕΛΚ, επαλήθευση. Για τη συμβαστική 51 γιατί ε, είναι λίγο αμφίβολο αυτό που βλέπω πέρας, αλλά υπάρχει πλειοψηφία, 25 προς 16 μια αποχή. Επίσης εγκρίνεται. Και άρα περνάμε κατευθείαν στην 143. Οι συνεισηγητές μας μόνοι τους κιόλας ε, ε μας προτείνουν την τροπολογία 142 πέρα κατά αποχές εγκρίνεται. 144 υπέρ κατά αποχές επαλήθευση. 144 ψηφίστε, ψηφίστε, ψηφίστε. Πέρας, 23 προς 18 εγκρίνεται. Και πάλι το, η, μια τροπολογία 145 των δύο συνεισηγητών υπέρ. Ε, το έλκο δεν το δαχτυλάκι, υπέρ είναι. Επαλήθευση. Υπέρ, όλοι είναι υπέρ. Εκτός από αυτούς που είναι κατά. Ποιος είναι κατά τις 145 κανένας. Α, ζητώ συγγνώμη. Αποχές. Μία. Εγκρίθηκε. 146 καταστροφική τροπολογία. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Οι συνεισηγητές μας προτείνουν την 147 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Η πράσινη την 149 υπέρ κατά αποχές νομίζω ότι υπάρχει ψηφία αλλά στο εξακριβώσουμε για την 149 ψηφίζουμε ηλεκτρονικά ψηφίστε κάποιοι μιλάνε υγ, άλλοι με κάποιοι μιλάνε και δεν ψηφίζουν πέρας 26 προς 15 μία αποχή το μηχάνημα, σας πληροφορώ, μας λέει ότι υπάρχει ένας περίφημος πράσινος προτού καν αρχίσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Απίστευτο. Κάποια μεγάλη πολυεθνική κρύβεται ε, από πίσω. Νομίζω ότι το ΕΛΚ, ε, λέει ο κύριος ε, ο Μάρκους, κυκλοφορείται αυτές τις φήμες. 150 των συνσηγητών υπέρ κατά αποχές Εγκρίνεται. 153. Γκουε υπέρ. Κατά. Αποχές. Έλεγχος. Υπάρχουν ε, περίεργες ε, συμμαχίες για την 153. Πέρασε 21 προς 20 με αποχή εγκρίθηκε. 155 η FTD υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 154 τώρα τη ανελίζει υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίθηκε. 156 πράσινη υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 157 η FTD υπέρ. Αποχές. Απορρίπτεται. Συμβαστική 52. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 160 περνά μόνο. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 161 της γκου υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. 162. Η FTD. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 163 Μάρκους Φέμπερ υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Συμβαστική 53 υπέρ κατά αποχές εγκρίθηκε. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ε, να τις ψηφίσουμε όλες μαζί, τις τελευταίες τροπολογίες. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 είναι ήδη οι συντάκτες. Ε, μπορούμε να τις ψηφίσουμε πολύ ωραία υπέρ. Κατά. Αποχές. Βλέπω μία πνοή, ένα κύμα ενθουσιασμού. Εκπληκτικό. Με ονομαστική ψηφοφορία. Τελική ονομαστική ψηφοφορία. Bon. Euh, oui. Alors, pardon, pardon. Avant de donner le résultat du vote. Πριν δούμε το αποτέλεσμα, η Γκουε μας ζητάει το λόγο ε, εξήγηση ψήφου. Ευχαριστώ. Θα ήθελα ε, να γραφτεί στα πρακτικά ότι από πλευράς διαφόρων βουλευτών της ομάδας GUE NGL θα θέλαμε να σημειωθεί η άποψη της μειοψηφίας, της δικής μας μειοψηφίας για αυτό το θέμα που εστάλει και στους συζητητές και στη γραμματεία. Με συγχωρείτε λέει ο πρόεδρος, θα έπρεπε να σας έχω δώσει το λόγο πριν από την τελική ψηφοφορία. Και από αυτή την ενημέρωση, αν θέλετε να αλλάξετε την ψήφο σας μπορείτε να το κάνετε, αλλιώς η ψηφοφορία. Οπότε 25 υπέρ, 6 κατά, 9 αποχές. Εγκρίνεται η έκθεση Συγχαρητήρια στους δύο συνεισηγητές μας. Ευχαριστώ και τους Κιώδης. Ευχαριστώ όσους συμμετείχαν στις εργασίες και στην ψήφο. Περιμένετε, περιμένετε, δεν έχει λήξει η συνεδρίαση. Υπενθυμίζω ότι η διαβούλευση των εγγράφων τις ομάδες για τον κώδικα διοντολογίας εξακολουθεί να είναι δυνατή η αίθουσα είναι ανοιχτή και όλες ε, οι τυπικές διαδικασίες είναι ενισχύ μέχρι τις 28 τρέχοντος Ιουνίου λίγη συνεδρίαση.